κατάσταση της συγκέντρωσης γεωργικών γεών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το πώς θα διευκολυνθεί η πρόσβαση των γεωργών στη γη. Επαναλαμβάνω, πρόκειται για σύντομη παρουσίαση της έκθεσης κυρίας Νόιχλ. Θα δώσω τώρα το λόγο πρώτα στην εισηγήτρια, την κυρία Μαρία Νόιχλ. Αξιότιμη κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι, λίγα λεπτά πριν χτυπήσει 12 το ρολόι, αλλά παρόλα αυτά έχουμε ένα ακόμα σημαντικό θέμα στην ημερησιά διάταξη. Μπορεί να ε, συζητάμε πολλά, όμως ε, χωρίς να το παρατηρούμε πίσω μας ε, όλο και περισσότερη γεωργική γη συγκεντρώνεται στα χέρια ολίγων σε γεωργικούς ομίλους. Ε, ή άλλους ομίλους. Το 3% των εταιριών ελέγχουν ήδη το 5% των γεωργικών γεών στην Ευρώπη και μόνο αυτό το νούμερο νομίζω ότι αρκεί για να καταλάβουμε τις ανησυχητικές διαστάσεις του φαινομένου. Επέκθεση λοιπόν πρωτοβουλία για τη συγκέντρωση γης ε, στην Ευρώπη είναι σημαντικό. Και το δεύτερο τμήμα της έκθεσης είναι πώς μπορούμε να διευκολύνουμε την πρόσβαση στη γη για τους αγρότες. Θα ήθελα πάρα πολύ σύντομα να αναφέρω οκτώ σημεία τα οποία Αναφέρουμε και στην έκθεση και βέβαια θέλω να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε όλοι τους σκιώδεις εισηγητές. Αναφέρουμε στην έκθεση ξεκάθαρα ότι δεν είναι ένα οποιοδήποτε αγαθό ε, διότι δεν είναι άπειρο, είναι πεπερασμένο, δεν μπορεί να πολλαπλασιαστεί, δεν είναι ένα εμπορικό αγαθό σαν οποιοδήποτε άλλο. Εμείς ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να κάνει κάτι ώστε να ε, φροντίσει την εφαρμογή των ε, κατευθυντήριων γραμμών και θα πρέπει να στηριχθούν τα κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά ε, την αγοραπολισία γεωργικών γεών. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Πρέπει να σταματήσει η αγοραπολισία και μέσω άλλων, σε άλλα κράτη και σε τρίτα βέβαια. Και αυτό το οποίο απαιτούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι από τα κεντρικά σημεία, απαιτούμε να συντάξει έναν κατάλογο κριτηρίων που θα αναφέρει συγκεκριμένα κριτήρια. Πώς μπορούν δηλαδή τα κράτη-μέλη ε, χωρίς διακρίσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση να βοηθήσουν να αποτραπεί ε, η αγοραπολισία γεών. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος απάτης και διαφθοράς. Θέλουμε επίσης ε, να υπάρχει ένα παρατηρητήριο για την αγορά γεωργικής γης, ε, ώστε να υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία και να μπορεί να δρά μετά αυτό το παρατηρητήριο και να βλέπουμε επίσης και πώς ε, προχωρά ε, και προοδεύει η συγκέντρωση γης στην Ευρώπη. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι αναφέρουμε συγκεκριμένους στόχους για την Ευρώπη, γιατί σε ό,τι αφορά τη διασπορά της έγκυας ιδιοκτησίας, αυτό δεν είναι μια σοσιαλιστική ε, ιδέα. Είναι μια ουσιώδης αρχή την κοινωνική οικονομία, είναι κάτι καλό και πρέπει να υποστηριχθεί. Επίσης επαναλαμβάνουμε και είναι και αυτό ένα σημαντικό σημείο αναφέρουμε τα βασικά ε, στοιχεία της ε, γεωργικής πολιτικής και του γεωργικού μοντέλου στην Ευρώπη, που ουσιαστικά ε, δεν βασίζεται μόνο στην παραγωγή μοντέλων, που φυσικά και είναι ένας απόλυτα θεμητός στόχος, αλλά ο βασικός στόχος της ΚΑΠΑ είναι η προστασία του περιβάλλοντος, της βιοπικιλότητας των εδαφών και των υδάτων. Αυτό είναι το ευρωπαϊκό γεωργικό μοντέλο. Αυτό θέλουμε να το υποστηρίξουμε και αυτό σημαίνει ότι θέλουμε να έχουμε όχι λίγες αλλά πάρα πολλές γεωργικές εκμεταλλεύσεις ε, διαφορετικές ε, και όχι μόνο λίγες. Επίσης ότι αφορά τη συγκέντρωση του χρήματος όλο και λιγότερα χέρια αυτό οδηγεί στα ίδια αποτελέσματα που οδηγεί και η συγκέντρωση της γεωργικής γης όλο και λιγότερα χέρια. Έχει τα ίδια μενεκτήματα στην έκθεση επίσης αναφέρουμε ξεκάθαρα και τη μελλοντική κατεύθυνση που θα πρέπει να έχει η πολιτική γεωργίας. Αν πιστεύουμε ότι θα πρέπει να έχουμε μόνο μία ενίσχυση ε, στρεματική, ε, καταλαβαίνουμε ότι αυτό δεν μπορεί να είναι βιώσιμο γιατί οδηγεί σε δυσανάλογη στήριξη των μεγάλων εκμεταλλεύσεων και ευνοεί τη συγκέντρωση της ε, γεωργικής γης. Έχουμε λοιπόν πολλά, πολλή δουλειά να κάνουμε ακόμα. Αγαπητοί συνάδελφοι, φυσικά το μπαλάκι τώρα είναι ξεκάθαρα στη, ε, στο γήπεδο της Κομισιόν και στο γήπεδο των κρατών μελών. Εμείς ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάναμε ό,τι μπορούσαμε και με ότι αύριο θα ψηφίσουμε με συντριπτική πλειοψηφία την έκθεση αυτή γιατί νομίζω ότι ε, σπάνια απαντά κανείς τέτοια ομοφωνία ε, όπως αυτή την περίπτωση όπου μιλάμε για ανάγκη τερματισμού της συγκέντρωσης γεωργικής γης. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Έχουν περάσει τα μεσάνυχτα. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, έχουμε περάσει ήδη στην Πέμπτη. Τι να κάνουμε, έτσι ήρθαν τα πράγματα. Μετά την εισηγήτρια θα περάσουμε στη διαδικασία Catch the Eye. Πέντε λεπτά για τη διαδικασία αυτή. Πάνω από δέκα συνάδελφοι ζήτησαν το λόγο, αλλά πρέπει να βρούμε μία λύση. Θα δώσω το λόγο μόνο σε όσους δεν το ζήτησαν ακόμη. Αυτοί έχουν προτίμηση. Θα ξεκινήσουμε από την κυρία Σένερα Ροντρίγκες. Είναι παρούσα η κυρία Ροντρίγε. Μάλιστα, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η συγκέντρωση γεών είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δυσκολεύει την εγκατάσταση ε, στην ύπεθρο των νέων ή των ακτιμώνων και μάλιστα εμποδίζει τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις να αναπτυχθούν. Πολλοί είναι οι λόγοι. Κερδοσκοπία, απαλωτρίωση για εξορρυκτικές ε, ή άλλες δραστηριότητες. Τελικά το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σφυράν κλέφτηκα, θελοτυφλούν όταν οι κυβερνήσεις ε, επιτρέπουν τέτοια διαδικασία και τη μη γεωρική χρήση των γεών αυτών. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε την προστασία των γεωρικών γεών με μέτρα που θα διασφαλίζουν και θα δίνουν προτεραιότητα στην κοινωνική λειτουργία της παραγωγής τροφίμων και θα προβλέψουν μηχανισμούς για να σταματήσει αυτή η συγκέντρωση και η, η φαρπαγή των γεών. Επίσης θα επιτρέψουμε σε νέους, σε γυναίκες ή σε οποιοδήποτε θέλει να ασκήσει γεωρική δραστηριότητα να έχει πρόσβαση στις γεωρικές γεές. Ευχαριστώ. Η κυρία Μαρία Χόιμπους κυρια μαρια χοιμπου εχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Μαρία Νόιχελ, την εισηγήτρια, η οποία πραγματικά ε, δούλεψε πάρα πολύ ανοιχτά, χωρίς να αποκλείσει κανέναν. Μπορέσαμε να καταλήξουμε σε καλούς συμβιβασμούς. Έγινε η προσπάθεια προς αυτό. Πραγματικά Υπάρχει αυτό το πρόβλημα της συγκέντρωσης ε, των ε, γεών, αυτό είναι διαμφισβήτητο, όπως είναι αδιαμφισβήτητο ότι και η εθνική νομοθεσία ε, δεν κάνει ό,τι μπορεί για να αποτρέψει τα φαινόμενα αυτά. Το θέμα είναι ε, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Παραδείγματο χάρη με τη γεωρική πολιτική, η περιφερειακή ανάπτυξη, το είπαμε, πολιτική, οικονομική, ε, δημοσιονομική ε, που επηρεάζει, επενδύσεις όλα αυτά. Έχουμε κερδοσκοπία με τη γη που αντιμετωπίζεται ως επενδυτικό αγαθό ε, τελικά και γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης. Όμως ε, η γη είναι κάτι πολύτιμο, όχι μόνο για μας τους αγρότες που παράγουμε για αυτή την εσωτερική αγορά μπορούμε και πρέπει να αγοράζουμε τα, και να πουλούμε τα πρώτα μας στην ίδια αυτή εσωτερική αγορά. Και θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες κατευθυντήριες γραμμές που να είναι η, αφετηρία για την προστασία των βασικών προϋποθέσεων ε, για την επιβίωση όχι μόνο των αγροτών ε, και αγροτισών της Ευρώπης αλλά και για όλους, την επιβίωση όλων των συμπολιτών μας. Ευχαριστώ κύριε Μορβάη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω ότι η έκθεση αυτή έχει πολύ μεγάλη σημασία. Είναι μια ιστορική έκθεση. η υγιής δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι η εγγύηση για την επιβίωση των ανθρώπων και είναι φυσικά ο τρόπος παραγωγής προϊόντων που είναι απαραίτητα για όλο τον κόσμο. Συνεπώς λοιπόν θα πρέπει να δώσουμε πάρα πολύ μεγάλο βάρος, δεν θα πρέπει εδώ να αφήσουμε το μεγάλο κεφάλαιο να δημιουργήσει υπερσυγκεντρώσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση φοβάμαι ότι αυτό προωθεί και γι' αυτό θα ήθελα να ζητήσω από τον Επίτροπε Έτιγκερ και την εισηγήτρια αν μπορούν να καταλήξουν επιτέλους τα σωστά συμπεράσματα ότι δηλαδή η ελεύθερη ε, διακίνηση των κεφαλαίων είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με διαφορετικό τρόπο. Στη συνθήκη ένταξης της Ουγγαρίας θα πρέπει να υπάρξουν αλλαγές και η γης δεν θα πρέπει να θεωρείται κάτι το οποίο μπορεί να αγοράζεται και να πωλείται σαν οδήποτε άλλο προϊόν η κυρία Λόπες Μπερμέχο. Ευχαριστώ. λοιπόν που αυτή η συζήτηση για την πρόσβαση στη γη γίνεται στα μεσάνυχτα, διότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα, κομβικό για την Ευρωπαϊκή Γεωργική Πολιτική στη χώρα μου, την Ισπανία έχουμε να αντιμετωπίσουμε και την εγκατάλειψη αγροτεμαχίων ε, που είναι πολύ κατακαιρματισμένα αυτά τα μετά για να, ε, τεμάχια για να είμαστε αποτελεσματικοί ενώ οι δύο χώρες του Νότου κάποιοι μεγάλοι γεωκτήμονες συγκεντρώνουν στα χέρια τους ε, τα μεγάλες γεωργικές επιφάνειες εκμεταλλευόμενοι τους εργάτες και πρέπει να πούμε πόσο μεγάλη σημασία έχουν οι πολιτικές σχεδιασμού, οι τράπεζες γεών, οι δημόσιες πιστώσεις, τα δάνεια και η ανάγκη να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της συγκέντρωσης, συγκέντρωσης γης. Ε, η γη ουσιαστικά ε, πρέπει να ε, ζει αυτόν που την δουλεύει και πραγματικά θα πρέπει να φροντίσουμε να επιβιώσουν οι μικρές αγροτικές εκμεταλλεύσεις και οικογενειακές εκμεταλλεύσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πέντε λεπτά προβλεπόταν για το ΚΑΤΣΔΙ. Εξαντλήσαμε το πεντάλεπτο. Ε, ζητώ συγγνώμη από τους υπόλοιπους ε, συναδέλφους που δυστυχώς δεν πρόλαβαν να λάβουν το λόγο. Αλλά αυτό είναι το πρόγραμμά μας και πρέπει να το τηρήσουμε. Ο Επίτροπος Έτιγκερ τώρα έχει το λόγο, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, Αξιότιμες κυρίε και κύριοι βουλευτές, θέλω να ευχαριστήσω την βουλευτή κυρία Νόιχελ καθώς και τους συναδέλφους της οι οποίοι ε, συνέταξαν την έκθεση αυτή είναι μια πολύ σημαντική ανάλυση για την ιδιοκτησία και την χρήση ε, των γεωργικών γεών στην Ευρώπη ε, αυτό που γίνεται στην έκθεση και έτσι πρέπει να πω ότι πραγματικά και εμείς ε, καταγράφουμε και την κατανομή ε, των γεών από πλευράς ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπής και σίγουρα υπάρχουν σημαντικές λειτουργίες πρέπει να υπόψη και σημαντικές επιπτώσεις σε ό,τι αφορά την ιδιοκτησία των γεωργικών γεών. βλέπουμε τι κάνουν, ποια είναι η σταθεροποιητική αξία και οι γνώσει ε, και η ευθύνη είναι σημαντική για την Ευρωπαϊκή Ένωση εν γέννη, για τις περιφέρειες. Ε, όλα αυτά τα σημειώνουμε και νομίζω ότι μπορούμε με αυτές τις παρατηρήσεις ε, να διαμορφώσουμε αναλόγως και τη μελλοντική γεωργική πολιτική Φυσικά ε, έχουμε υπόψη ε, τους ε, νέους αγρότες, θέλουμε να παραμείνουν στο επάγγελμα αυτό και οι επόμενες γενιές, θέλουμε να τους δώσουμε μία προοπτική και σε ό,τι αφορά την ε, συγκέντρωση και σε ό,τι αφορά την ε, βιομηχανία τροφίμων ε, θέλουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε να προωθήσουμε την οικονομία της υπαίθρου των αγροτικών περιοχών. Βέβαια εδώ βλέπουμε μια σύγκρουση στόχων αν θέλετε. Από τη μία φυσικά και υπάρχει στο ευρωπαϊκό δίκαιο η αρχή της επένδυσης που κατοχυρώνεται. Οποιοςδήποτε μικρός μεγάλος μπορεί επιτρέπεται να επενδύει σε κάποια αγαθά ως Ευρωπαίος πολίτης στη δική του τη γη, ε, στη δική του χώρα, σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα ε, ή σε κάποια τρίτη. Υπάρχει αυτή η ελευθερία. Και από την άλλη πλευρά τα κράτη-μέλη έχουν τη δυνατότητα να ε, λάβουν μέτρα κατά της συγκέντρωσης και δι της κερδοσκοπίας της γης και να φροντίσουν να προστατεύσουν, να βάλουν σε ένα καθεστώς προστασίας ε, τις ε, γεωργικές γης. Ε, τα τελευταία χρόνια είχαμε επαφές και διαβουλεύσεις με τα κρατημέλη και με τις περιφέρειες και προσπαθήσαμε να δούμε πώς μπορούν να λειτουργήσουν συγκεκριμένα μέτρα προστασίας και περιορισμού Και είδαμε επίση πως κάποια μέτρα μπορεί άμεσα ή έμεσα να συνιστούν διακριτική μεταχείριση. Είχαμε τις επαφέ με τα κράτη-μέλη. Εμείς θα συνεχίσουμε αυτέ τις επαφέ με τα κράτη-μέλη έχοντας ως βάση και το δικό σας έγγραφο, τη δική σας έκθεση. Θα συνεχίσουμε τις συζητήσει και με εσάς αλλά και με τα κράτη-μέλη και εγώ και οι υπόλοιποι αρμόδια για τον προπολογισμό επίτροποι που θα ασχοληθούμε στο μέλλον με τη μεταρρύθμιση και τη ε, κοινή γεωργική πολιτική, ε, θα λάβουμε υπόψη μα ε, τι συστάσει. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Ολοκληρώσαμε και το θέμα αυτό.